Okay. So, good morning, colleagues. Uh, welcome to our econ... Καλημέρα. Αντικαθιστώ τον κύριο Γκουαλτιέρη σήμερα, λέει ο κύριο Χάιε. Σήμερα το πρωί ξεκινάμε με δύο επιτροπές και επειδή θα έχουμε περισσότερους ε, ευρωβουλευτές, γι' αυτό καθόμαστε έτσι. Λοιπόν, να δούμε την ημερήσια διάταξη. Το σημείο 2 είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Συμφωνούμε? Ωραία, συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων που έχετε στη σφαγέλου σας. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε. Ωραία. Δεν έχω ανακοινώσεις στο σημείο 4. Σημείο 5. Έγκριση του σχέδιο χρονοδιαγράμματος Ιούλιο με Δεκέμβριο 2019 για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο σημείο 6 το οποίο είναι η ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσει. Το σημείο 6 λοιπόν έχω να κάνω διάφορε ανακοινώσει. Πρώτον, πρόκειται για τη διασυνοριακή κατανομή των κονδυλίων 5 ε, Φεβρουαρίου. Δεύτερο τρεμερή διάλογο ε, λοιπόν έγινε στι 5 Φεβρουαρίου και καταφέραμε να καταλήξουμε όσον αφορά τα διάφορα πολιτικά σημεία, κυρίως για το σημείο που έχει να κάνει με την αποκοινοποίηση των επενδυτικών ε, ταμείων για εναλλακτικά ταμεία και για να επεκταθεί η προθεσμία σχετικά με τα PRIPS, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ταμεία usage, ο ΣΕΚΑ. Ε, προβλέπω λοιπόν ότι θα συνεχίσουμε τις επόμενες εβδομάδες και ο στόχος είναι να εγκρίνουμε στην Ολομέλεια το τελικό κείμενο στη δεύτερη Ολομέλεια του Απριλίου. Ερχόμαστε τώρα στο ΕΜΙΡ 1 REFIT. Ο τριμερής διάλογος 5 Φεβρουαρίου έγινε ο τελικός τριμερής διάλογος της 5 Φεβρουαρίου και οι συνομοθέτες κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής για το φάκελο αυτό. Ε, υπήρξε συμβασμός όσο αφορά για τη διάρκεια της εξαίρεσης για τα clearing obligations όσον αφορά τις δαξιδιωτικά και το κείμενο που προτείνεται θα οριστικοποιηθεί σε τεχνικό επίπεδο και θα υπάρξει τις επόμενες εβδομάδες μια επόμενη συνάντηση σε επίπεδο Επιτροπής. Τριμερής διάλογος τώρα για τον κανονισμό όσον αφορά για την ε, ε, δημοσιοποίηση σχετικά με τις βιώσιμες επενδύσεις, 12 Φεβρουαρίου. Οι διαπραγματευτικέ ομάδες κατέφεραν να καταλήξουν σε ε, συμβαστικές προτάσεις πάνω στο κείμενο όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης σε διάφορα επίπεδα και για την εξωτερήκευση του, των πτυχών του ECG. Ο επόμενο τριμερή διάλογο θα γίνει στι 27 Φεβρουαρίου. Και όσον αφορά τώρα για τον τριμερή διάλογο 6 και 12 Φεβρουαρίου, όσον αφορά τι επενδυτικέ εταιρείε, έγιναν δύο τριμερεί διάλογοι και προτάθηκε ένα πακέτο και υπάρχουν καταρχήν συμβασμοί για διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν ε, με τις αμοιβέ, τα bonus cap, την ε, ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, τις απαιτήσει ρευστότητα, περιβάλλον κοινωνικά κλπ. Χρειάζονται πάντως παραπετέρω συζητήσεις για να καταλήξουμε για αυτά τα θέματα, κυρίως για το πεδίο εφαρμογή του IFR, τους ε, κανόνες ισοτιμίας, τις κεφαλαϊκές απαιτήσει στους παράγοντες K, και ναι, επόμενο τριμερή διάλογο είναι 26 Φεβρουαρίου. Τώρα, ε, καλυμμένα ομόλογα. ομόλογα. διάλογος 13 Φεβρουαρίου. Έγινε ο τρίτος τριμερή διάλογος τότε και διάφορα θέματα όπω είναι οι δομέ ληκτικότητα, όπω είναι μεταβατικά μέτρα ισοτιμίε με τρίτε χώρε που δεν είχαν συζητηθεί προηγουμένω. συζητήθηκαν αυτή τη φορά. Παρετέρω συζήτηση για τα καλυμμένα περιουσιακά στοιχεία ε, έγινε και βοήθησε να υπάρξει παρατέρω κατανόηση μεταξύ των δύο συνομοθετών. Θα υπάρξει επόμενο τριμερή διάλογο την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι έχω καταλάβει, και θα γίνουν και τεχνικέ ε, συναντήσει. Ε, τριμερή διάλογο για τα κριτήρια, benchmarks. Τρίτο τριμερή διάλογο έγινε στο Στρασβούργο 13 Φεβρουαρίου και συζήτησαν οι διαπραγματευτικέ ομάδε για τα μεταβατικά κριτήρια και για τα κριτήρια ευθυγράμμιση με το Παρίσι. Ε, τα κριτήρια για το κλίμα θα πρέπει να αποτελούνται από επιλεγμένα κριτήρια βάσει της διαδρομής ε, αποφυγής του άνθρακα. Ο επόμενος τριμερής διάλογος προβλέπεται για τις 25 Φεβρουαρίου. Έρχομαι τώρα στο ESFS και εδώ έγινε τριμερής διάλογος. Ο πρώτος 14 Φεβρουαρίου. Όλες οι πλευρές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να καλύψουν όλη την αναθεώρηση της διαπραγματεύσης. Επετέχθη πρόοδος για τις πτυχές ε, του ξεπλήματος χρήματος, νομιμοποίησης παράνομου χρήματος και επιτεύθηκε και κάποια συμφωνία όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή. Η επόμενη συνάντηση προβλέπεται για την 21η Φεβρουαρίου και εκεί θα συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της νομοποίησης παράνομου χρήματος και βάσει των άρθρων 1 με 38 της ΣΥΜΠΙΑ. Ε, χτες έγινε και ο τέταρτος του διάλογος για το ΕΜΗΡΔΙΟ 2.2 σχετικά για τη διακυβέρνηση, για τα δικαιώματα ψήφου, για θέματα που έχουν να κάνουν με την εποπτεία των CCP's, ε, την Εποπτική Επιτροπή και την ανάμειξη της ΕΣΜΑ στην λήψη αποφάσεων. Και επίσης όσον αφορά για τρίτες χώρες κοινέ διατάξεις είναι η διαδικασία για την άρνηση της αναγνώρισης και την ανάμειξη των κεντρικών τραπεζών. Επιπλέον έγινε και μια πρώτη άτυπη συνάντηση και συζήτηση για την τροπολογία στο άρθρο 22 για το καθεστώς CCB. Πρόκειται να υπάρξει επίσημος τριμερής διάλογος χωριστά τις επόμενες εβδομάδες. Αυτά και ερχόμαστε τώρα στο σημείο 7. Μάλλον σας είπα λοιπόν, αυτή ήταν η ενημέρωση για τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις και τώρα ερχόμαστε στο σημείο 7, το οποίο έχει να κάνει με τον έλεγχο των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων. Πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε όσον αφορά τα PRIPS συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασισμένα σε ασφαλίσεις. Πρόκειται και για τα εφαρμοστικά μέτρα, όπως ξέρετε. Κάθε φορά που αρχίζει ένα, ένας νέος κύκλος εποπτείας, και αυτός είναι ο 42ος η Επιτροπή Εκόνο δίνει μεγάλη σημασία στην ε, πραγματική και αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών αυτών ε, αρμοδιοτήτων. Σήμερα λοιπόν θα επικεντρωθούμε στην κατάσταση πραγμάτων για τα εκτελεστικά μέτρα όσον αφορά τα PRIPS. Υπάρχουν τροπολογίες από την ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ και κάποιες διατάξεις πριπς ήδη συζητήθηκαν στις ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις επί των νομοθετικών προτάσεων για τη διευκόλυνση της κατανομής των επενδυτικών ταμείων διασυνοριακά. Επίσης, όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση, η κοινή αρχή της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής ε, της Εποπτικής ξεκίνησε διαβουλεύσεις για την κατεξοδότηση πράξη πρίψη και επίσης όσον αφορά τα έγγραφα βασικών πληροφοριών. Οι τελευταίες συστάσεις αρχές Φεβρουαρίου λέ, καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα και λένε ότι αυτή η διαβούλευση θα έπρεπε να επεκταθεί και να υπάρξει και μια δημοσιοποίηση των πληροφοριών όσον αφορά τις επιδόσεις. Θα δώσω το λόγο στον Γκάμπριελ Μπερναντίνο που είναι ο πρόεδρος της ΕΙΟΠΑ και είναι και πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Εποπτικών Αρχών και τον Σβέν Κέντνερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μιλήσουν στο σώμα ο κύριος Μπερναντίνο ίσως πρώτα και μετά θα υπάρξει και συζήτηση βέβαια. Οπότε κύριε Μπερναντίνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε και χαιρετίζω φυσικά τους ευρωβουλευτές. Όπως είπατε είμαι εδώ ως πρόεδρος της Μεκτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και θα σας μιλήσω για τα πρίψ. Και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω για το έργο μας όσον αφορά τις κατεξοδότηση πράξης για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν τα πρίψ. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπογραμμίσω ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στα έγγραφα βασικών πληροφοριών γιατί έτσι βελτιώνεται η διαφάνεια των ε, επενδυτικών προϊόντων μέσω τυποποιημένου εντύπου δημοσιοποίησης. Εμείς θέλουμε πάρα πολύ να στηρίξουμε την αποτελεσματική και με σύγκληση εφαρμογή και υλοποίηση των κανόνων όσον αφορά τα διάφορα προϊόντα που κυκλοφορούν πολύ διαφορετικά σε διάφορες χώρες να διευκολυθούν αυτοί που παράγουν τα πρίψα αλλά και κυρίως οι καταναλωτές, κυρίως αυτοί που δρούν διασυνοριακά. Επίση, θέλουμε να θεωρήσουμε του υπάρχοντε κανόνε εκεί που αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται εξίσου καλά σε παντό είδου πρίψη. Και είναι φυσιολογικό οι κανόνε που είναι βέβαια περίπλοκοι, να πρέπει να διευκρινίζονται και να αναθεωρούνται βάσει της εμπειρίας που συλλέγουμε και βάσει του τι βλέπουμε ότι λειτουργεί καλά και τι λειτουργεί λιγότερο καλά. Καταλαβαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν θέσει κάποιες ανησυχίες για διάφορες πτυχές. Τα εξετάζουμε όλα αυτά και εξετάζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Σε μερικέ περιπτώσει μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε ερωτήσει και απαντήσει για να απαντήσουμε διάφορα τεχνικά ζητήματα. Αποφασίσαμε όμω το φθινόπωρο που μα πέρασε ότι το καλύτερο που είχαμε να κάνουμε για πολλά αυτά τα ζητήματα ήταν να προτείνουμε κάποιε στοχευμένε τροπολογίε στον καταξιοδότηση κανονισμό πριψ. Ξεκινήσαμε λοιπόν την διαβούλευση τον Εύρεο που μα πέρασε και επικεντρωθήκαμε στι υποθέσει εργασία σχετικά με τι επιδόσει. Γιατί σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω εκεί. Αυτό αποτελεί μέρος βέβαια των βασικών γράφων και έχουμε προτείνει αλλαγές και στην ε, διαβούλευση για να αποφύγουμε ε, επικάλυψη των δημοσιοποιήσεων που γίνονται ανάμεσα στα ΠΡΙΠΣ και τους ΣΟΣΕΚΑ. Τώρα θέλω να συνοψίσω σύντομα ποια είναι τα θέματα τα οποία, οποία κατέληξε η διαβούλευση. Πρώτα απ' όλα υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόνων ότι οι υποθέσεις εργασίας για τι επιδόσει δεν θα πρέπει να θεωρηθούν σαν προβλέψει. Υπάρχει ο κίνδυνο οι καταναλωτέ να νομίζουν ότι πρόκειται για προβλέψει. Οι ενδιαφερόμενοι επίση εξέφρασαν ανησυχίε για το σημερινό οικονομικό περιβάλλον ότι μπορεί να οδηγήσει στο να μην ε, βλέπουμε την, τις προσδοκίες που υπάρχουν από τις αγορές και τελικά να καταλήξουν αυτές να είναι προς τα κάτω. Οι προτάσεις οι μας στηρίζουν αυτές τις ανησυχίες. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις όσον αφορά την μεθοδολογία του σεναρίου βάση επιδόσεων και γι' αυτό προτείνεται να αναλύσουμε περισσότερο το θέμα. Για διάφορα πρίψη, όπως είναι η ενεργητική διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, ε, πολλές οργανώσεις καταναλωτών έχουν την άποψη ότι τα πρίψ τον πρίψ η ε, παρελθούσα επίδοση είναι το καλύτερο που χρειάζονται για να μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Επίσης η διαβούλευση ε, έδωσε διάφορες απαντήσεις και όσον αφορά τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τη σημασία της αναθεώρησης της γνωστοποίησης του κόστους. Έτσι λοιπόν, όταν αποφασίζουμε για τις τελικές μας συστάσεις, λαμβάνουμε υπόψη μας όλα αυτά και θα συνεχίσουμε μέχρι το 2021 γιατί αποφασίσαμε την αναβολή της εφαρμογής του ΚΙΤ στους ΟΣΕΚΑ. Επίσης, σκεφτήκαμε ότι δεν πρέπει να βάλουμε πολύ στενές, πολύ συγκεκριμένες τροπολογίες σε αυτό το στάδιο, αλλά ότι θα πρέπει να μειωθεί ο κίνδυνος να υπάρξουν παρερμηνίες στα σενάρια σχετικά με τις τρέχουσες επιδόσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε εκδώσει μια εποπτική ε, ενημέρωση για την προστασία των ιδιωτών επενδυτών. Και σε αυτό το στάδιο προτείνουμε να συμπεριλαμβάνουν αυτοί που φτιάχνουν τα πρίψη μια προειδοποίηση μέσα στο βασικό έγγραφο για να ενημερώνουν τους ιδιώτες επενδυτές ώστε αυτοί να γνωρίζουν τους περιορισμούς και τους κινδύνους. Τον Φεβρουάριο επίσης αποφασίσαμε ότι θα ξεκινήσουμε μια αναθεώρηση του κατεξοδότηση κανονισμού των πρίψη ήδη φέτος. Και τώρα θα τελειώσω με τα εξή θέματα. Πρώτο, θέλουμε να καλύψουμε θέματα επιδόσεων όπω επίση και γνωστοποίηση κόστου. Θα συμπεριλάβουμε μια αξιολόγηση για το κατά πόσο η μεθοδολογία του κόστου και η μείωση τη απόδοση είναι η σωστή προσέγγιση ή πρέπει να τροποποιηθεί. Επίση, θα καταλήξουμε σε ανάλυση για το βασικό έγγραφο και ε, ετησίως θα ενημερώνουμε για το κόστος και τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδυτικών προϊόντων. Θα επικεντρωθούμε επίσης σε τροπολογίες όσον αφορά τον καταξιδότηση κανονισμό πρίψ. Όμως, εκεί που το έργο μας δείχνει ότι αλλαγέ στα πρίψ επίπεδο 1 του κανονισμού αυτού δηλαδή χρειάζονται για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο επίπεδο 2, τότε θα συστήσουμε αλλαγές δεδομένου του μεγάλου πεδίου εφαρμογή του κανονισμού και να διασφαλίσουμε ότι το βασικό έγγραφο λειτουργεί ικανοποιητικά για όλα τα προϊόντα, προτείνουμε και διαφοροποίηση ανάλογα με τον τύπο των PRIPS. Ε, παρόλο βέβαια που θέλουμε να υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ των ε, προϊόντων υποκατάστασης. Τέλος, θέλουμε να κάνουμε και δοκιμές με τους καταναλωτές και όσον αφορά το σημερινό βασικό έγγραφο και όσον αφορά εναλλακτικές λύσεις. Θέλουμε να μείνουμε πολύ κοντά στους αρχικούς στόχους του κανονισμού, δηλαδή οι καταναλωτές να μπορούν πιο εύκολα να αντιληφθούν τις πληροφορίες που τους δίνουμε και να αποφεύγονται κίνδυνοι Επ' αυτού λοιπόν, καλωσορίζουμε φυσικά την συμβολή των Ευρωβουλευτών όσον αφορά τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα του βασικού εγγράφου έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τους καταναλωτές. Τέλος, καλωσορίζουμε την επιβεβαίωση ότι οι τροπολογίες στον κανονισμό PRIPS θα γίνουν φέτος όσον αφορά το θέμα της επικάλυψης της δημοσιοποίησης ανάμεσα στα PRIPS και του ΣΟΣΕΚΑ. Χρειάζονται κάποιες διορθώσεις για να ευθυγραμμιστεί ο ή κανονισμός και θα έχουμε νέες προτάσεις τις επόμενες εβδομάδες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το βασικό έγγραφο πρίψ θα λειτουργεί για όλα τα προϊόντα και για το ΣΟΣΕΚΑ. Έτσι, οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν μεταξύ επενδυτικών προϊόντων και θα μπορούν και ισότιμα να ε, λειτουργούν οι προμηθευτές των πρίψ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Περναρδίνο. επικεφαλής της Υποπτεύχους ε, αρχή. Παρακαλώ τώρα από τη Γενική Διεύθυνση μου. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Μας καλέσατε σήμερα να μιλήσουμε για τα επόμενα βήματα για τον κανονισμό ΠΡΕΠΣ. Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως τι πρόσφατες τροποποίησεις ε, στο χρονοδιάγραμμα για τα PRIPS που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε τι απαραίτητε προσαρμογέ στο δεύτερο επίπεδο έτσι ώστε να έχουμε, να έχουμε καλύτερη οργάνωση. Θα ήθελα ωστόσο να τονίσω πως ο συνολικός στόχος μας θα πρέπει να παραμείνει πως τα PRIPS θα πρέπει να έχουν τις καλύτερες δυνατές ε, προδιαγραφές και για το χρήστη τους. Ο στόχος του κανονισμού λοιπόν, η διαφάνεια και η ε, δυνατότητα συνεργασίας, η διαλειτουργικότητα μεταξύ των επενδυτών παραμένει. Και έτσι, όταν πρέπει να καλυφθεί ένα τόσο ε, περίπλοκο προϊόν, με τόσες διαφορετικές ε, δηλαδή εκφάνσεις, είναι ακόμη πιο δύσκολο να εξασφανιστούν ε, οι στόχοι. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας κάνουμε ή να λησμονήσουμε το γενικό στόχο. Αντί για μια προσέγγιση σιλό, δηλαδή ενιαία σε ένα δημοσιονομικό κανονισμό, έχει ζητηθεί να κοιτάμε χωριστά τα προϊόντα και από την προοπτική των επενδυτών. Ακριβώς αυτό γίνεται με το PRIPS. Ας μην αμφισβητηθεί λοιπόν η αρχή τη συγκρισιμότητα ή το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Α εστιαστούμε καλύτερα στην αντιμετώπιση σε πρακτικού όρου των προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε. Και για μα τα επόμενα βήματα πρέπει να είναι τα εξή. 2019. Όλε οι προσπάθειε θα πρέπει να εστιαστούν στην επίλυση των προβλημάτων επίπεδου 2. Ανέφερε και ο κ. Μπερναρντίνο την έκφραση των συμπερασμάτων ύστερα από τι διαβουλεύσει και βεβαίως θα πρέπει οι εποπτικές αρχές να αναπτύξουν τις λύσεις ανάλογα με τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει. Ωστόσο, ένα από τα κύρια προβλήματα, από τα ζητήματα που μένουν, είναι τα πιθανά σενάρια επιδόσεων και οι λύσεις σχετικές με το έγγραφο ενημέρωσης ε, στο το KID δηλαδή. Έτσι λοιπόν πρέπει να, να λυθούν αυτά τα ζητήματα τώρα και το Κοινοβούλιο πρέπει να βοηθήσει στην ε, εξέβρεση ενός τρόπου. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να αποφύγουμε επανελειμμένους γύρους ε, διαπραγματεύσεων τύπου για τις αλλαγές δηλαδή στο επίπεδο 2 των ΠΡΙΠΣ, μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς ως Επιτροπή ώστε να έχουμε έτοιμα, έτοιμες προτάσεις πριν από το 2021. Μπορεί να γίνει αλλαγή στο RTS ώστε από ένα προϊόν με πολλαπλές επιλογές να προσαρμοστούμε στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει προβλεφθεί από το τριμερή διάλογο. Παράλληλα με τη δουλειά για το RTS θα γίνει και η ευρύτερη επισκόπηση του, των προτάσεων PRIPS, ενδεχομένων ε, και εξαιρέσεων επίσης, με βάση το USET. Και όταν γίνουν οι αλλαγές σε καταθέτουμε πρόταση με βάση την έκθεσή μας για αλλαγές στο πλαίσιο usage και με βάση βέβαια πάντα το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. για αδίποτε αλλαγή από το usage που θα, πρέπει να μετα... θα, εισαχθεί θα πρέπει να μεταφραστεί και σε εθνικό δίκαιο. Άρα για να τηρηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα πρέπει οι αλλαγές στο RTS ε, πρέπει να συμφωνηθούν και οι αλλαγές στο usage πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται του χρόνου. Σημαντικά στοιχεία λοιπόν για την συνολική αναθεώρηση των πρίψ επιπλέον. Θα έχουμε τα ζητήματα της εξέτασης, της έκθεσης, για να δοκιμάσουμε και την χρήση του νέου ε, εγγράφου ενημέρωσης, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινήσουμε νωρίτερα το έγγραφο αυτό, εφόσον πρόκειται να γίνουν κάποιες αλλαγές του χρόνου και στο έγγραφο ΚΙΤ αλλά για δίποτε αλλαγή στο RTS και συμφωνώ εδώ με τον Γκαμπριέλ Περναρντίνο πρώτα να δοκιμαστεί και βέβαια να υποστεί και τη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Όταν έχει δε γίνει και η τελική επισκόπηση των ΠΡΙΠΣ, θα πρέπει να κοιτάξουμε μια ευρύτερη προσέγγιση να ακολουθήσουμε και όχι μεμονωμένα το kit, το έγγραφο ενημέρωσης. Γιατί έχουν γίνει αρκετέ αλλαγέ τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο των ΠΡΙΠΣ, αλλά και στο από το MIFID και από το IDT που αφορούν του επενδυτέ. Άρα λοιπόν και τι πληροφορίες που του δίνονται. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς συνδυάζονται τα νομοθετήματα αυτά, πώς μπορεί να βελτιωθεί η απόδοσή τους στην πράξη, εάν αρκούν οι πληροφορίες για τον επενδυτή, εάν είναι υπερβολικά πολλές επαναλαμβανόμενε, εάν οι μεθοδολογίες έχουν μάλλον συνεργατική ή μάλλον αποκλίνουσα δράση και όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν μέσα στην αναθεώρηση Ευχαριστώ πολύ και τους δύο ομιλητές μας. Και περνώ τώρα στην ομάδα αντιπραγμάτευσης πρέπει. Κύριε Μπερές. Μπορεί να ξεκινήσει και μετά περιμένουμε και τους συναδέλφους. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ όντως ε, απαραίτητο όταν πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία μέσα στην εντολή την τρέχουσα τη βουλευτική περίοδο τρέχουσα να κοιτάξουμε το θέμα των πρίψ Βέβαια η Επιτροπή επεδίωξε να υπάρχει ένα μόνο πακέτο κατεξιότηση πράξεων. Με συνέπεια αυτό να πάει για εξέταση στο προσεχέ κοινοβούλιο. Όμω τώρα ξεκινάει η συζήτηση και γι' αυτό είναι και απαραίτητο και εμεί να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε ε, ατάκτως ερημένα θα σας τα πω, ε, διάφορα σημεία όμως, ε, για τον Σβέν Γκέντνερ καταρχάς, ο οποίος ε, ανέφερε και λυπή εν εξελίξη νομοθεσία ή νομοθετική αναθεώρηση, που μπορεί να έχει κάποια συνάφεια να επηρεάσει την, το κεφάλαιο πρίψη. Μπορεί να κατάλαβα λάθος, αλλά πάντως δεν άκουσα να μιλάει για το προσπέκτους. γιατί είναι ένα θέμα καυτό, είναι ένα θέμα το οποίο διαρκώς ε, διατυπώνω ως ερώτημα. Συγκεκριμένα, εάν ή πόσο το η συνοπτική εκδοχή του προσπέκτους μπορεί να εξομοιωθεί με ένα έγγραφο ενημέρωσης για τους επενδυτές, ένα kit, ή να το αντικαταστήσει κιόλας. Γιατί δεν έχουμε πολλά έγγραφα τα οποία μπορούν να δώσουν ε, αρκετά χρήσιμες πληροφορίες, αποκαλυπτικές πληροφορίες, ιδιαίτερα για το μικρό επενδυτή. Ενώ υποτίθεται ότι όλη αυτή η προσπάθεια για μια αγορά των κεφαλαίων, κεφαλαϊκή αγορά, έχει σαν νόημα την επέκτασή της πέραν των επαγγελματιών επενδυτών στους μικροεπενδυτές. Άρα χρειάζεται και η πλήρης ενημέρωση αλλά και η συγκρισιμότητα. Κρίσιμη σημασία σε αυτό και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Καθημερινά λαμβάνω επιστολές από διαχειριστές χαρτοφυλακίων, ε, συνταξιδοτικών ταμείων λοιπά που θέλουν ο καθένα να επικαλεστεί την ιδιαιτερότητα της δικής του περίπτωση. Αλλά πρέπει πάντα να διατηρούμε εμείς τη στόχευση, ως βουλευτέ δηλαδή, την αναζήτηση της συγκρισιμότητας στην πληροφόρηση. Κάτι άλλο, πολύ σημαντικό επίση, που πρέπει να λύσουμε είναι τα σενάρια επιδόσεων και κυρίως προηγουμένων επιδόσεων. Συναρπαστική συζήτηση. Μα παρέσυρε σε διαλόγους και ανταλλαγέ κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, αλλά συνεχίζεται. Και πάλι πρέπει να ανοίξουμε κάποια λύση. Άλλοι λένε μηδέν, άλλοι λένε αποκλείεται, άλλοι λένε πολύ λίγο. Εάν θέλουμε όμω να παρουσιάζουμε τι προηγούμενε επιδόσεις, τι έχετε εσεί να προτείνετε έτσι ώστε αυτό να μην είναι παραπλανητικό και να υπάρχει και η προειδοποίηση αυτή που θέλετε να περιλάβετε. Δεύτερον, δεν συμφωνώ, δεν συμφώνησα με τη γραμμή που ακολούθησε το Κοινοβούλιο για το KIT και το Use It, γιατί πρόκειται για άλλη μια χειρονομία προς τους διαχειριστές ε, χαρτοφυλακίων και στρατιωτικών ταμείων που δεν βλέπω να έχει καμία χρησιμότητα. Έτσι λοιπόν ελπίζω είτε οι εποπτικές αρχές είτε η Επιτροπή εν τέλει να ε, επιδείξουν επιμέλεια και αυστηρότητα έτσι ώστε να τηρηθούν ε, απόλυτος οι προδιαγραφές, να προχωρήσουμε ταχύτερα, ενδεχομένως και να κλείσουμε νωρίτερα από τη διετία, αν είναι δυνατόν αυτό. Γιατί οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν ε, σαν σήμα καταθέτουν σε αυτή την προσέγγιση. Ε, λοιπόν, εάν μπορούσαμε να προστατέψουμε αυτό το κομμάτι της αγοράς, ώστε να μην ξεφύγει από τον έλεγχο ή την υποχρέωση ενημέρωσης που είναι η... το KID. Και επίσης ε, θα ήθελα να μου πείτε τι είδου στοιχεία θεωρείτε ότι θα ήταν αρκετά ή επίσης τι είδου δοκιμές μπορούν να γίνονται σημαντικό κομμάτι των ε, διαπραγματεύσεων ε, και όπως είπα πρέπει να το συνδυάσουμε και με την μετάβαση στο προσπέκτους και με τη συγκρισιμότητα με το Uset και άλλα και επίσης κάτι που και πραγματικά εξοργίζομαι δεν έχει καθόλου αντιμετωπιστεί ήθελε ο νομοθέτης RTS έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση μέσα στο έγγραφο KIT για τα χαρακτηριστικά που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με τα κριτήρια OSG. Η Επιτροπή Αγρών αγοράζει και στο συγγνώμη για τον κύριο Γκέντνερ με τον οποίο είχαμε πάντα εξαίρετη συνεργασία, αλλά εδώ μιλάμε για απάτη διανοητική. Μας λέγατε ότι θα υπάρχει ταξονομία, αμέσως ταξονομία δεν ήρθε, ακόμα δεν υπάρχει, ταξινόμηση πες περιπτώσει, δεν είναι δυνατό να προχωρήσουμε έτσι, δεν είναι λογικό και ταυτόχρονα δεν συνάδει και με το πνεύμα ενός από τα μεγάλα επιτεύγματα της Επιτροπής μας που είναι τα συμπεράσματα της ομάδας ψηλοεπιπέδου, της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Άρα λοιπόν, αυτό που προγραμματίζεται ως kit για το τέλος του χρόνου πρέπει και το πετώ να περιλάβει και στοιχεία για τις προϋποθέσεις επίπεδου 1 αυτό προς την Επιτροπή αλλά και προς εκείνους που θεωρούν ότι δεν ανήκει στην εντολή τους και ούτω καθεξής. Υπάρχει υποχρέωση αποτελέσματος. Εδώ. Ευχαριστώ, Περβάς. Είσαι το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις σας. Πολλά, μένουν, πολλά είναι τα σημεία που πρέπει να συμφωνηθούν. Ξεκινώ με την ε, ευθυγράμμιση όλων αυτών των ε, υλικών ε, κανονισμών και υλικών τεκμηρίωσης που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση του καταναλωτή. Όλα τα διάφορα φυλάδια και προσπέκτους ουσιαστικά είναι ένα τέρας. Πράγματι, συμφωνώ και υπάρχουν και διάφορα άλλα ζητήματα στις διαδικασίες για την τεξονομία. Έχουν έρθει σε τέλμα, δηλαδή βρισκόμαστε σε κάποιο τέλμα. Μας είχε υποσχεθεί η Επιτροπή στην αρχή των διαπραγματεύσεων ότι θα κάνει μια προσπάθεια και εμείς ε, συμφωνήσαμε ολόψυχα ότι θα έχουμε το KID, το βασικό πληροφοριακό έγγραφο για τα πρίψε και ε, κατανοητή, απλή, εύληπτη πληροφορία. Αυτό θα ήταν το μοντέλο για όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών με δυνατότητες συγκρισιμότητας, μόνο που οι μετοχές θα ήταν κάτι το πιο επικίνδυνο ως επένδυση σε σχέση με άλλους χρηματοπιστωτικούς τίτλους. Σε κάθε περίπτωση το Κοινοβούλιο αυτό θέλει να προωθήσει τη διαφάνεια, την απλούστευση και ελπίζαμε ότι η Κομισιόν θα αρχίσει να ε, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Και πολλά άλλα πρέπει να βελτιωθούν, όχι μόνο το το βασικό πληροφοριακό έγγραφο για τα οι περασμένες επιδόσεις. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Δεν θα επισέλθω επί μακρόν γιατί ε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε μεταξύ μας. Όμως ε, ανησυχούμε και είμαστε επεπισμένοι για το γεγονός ότι οι περασμένες επιδόσεις δεν είναι σωστός τρόπος να ενημερώνεται ο καταναλωτής. Είναι παραπλανητικές και είναι μη αξιόπιστες. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δηλαδή για παραπλάνηση και απουσία αξιοπιστίας και θα πρέπει να το αποφύγουμε. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει μια προειδοποιητική σήμαση. Ε, αυτό υπάρχει ήδη, ότι οι παρελθούσες επιδόσεις δεν ε, σημαίνουν ότι το ίδιο θα ισχύσει ε, και για τη μελλοντική έκβαση της σημερινής ε, επένδυσης. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σήμαση, αλλά τότε γιατί, βάζουμε, γιατί βάζουν οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πληροφορίες για τις παρελθούσες επιδόσεις όταν προειδοποιούν ότι αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι αξιόπιστη. Δεν έχει πολύ νόημα αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί δεν αρκεί απλά αυτή η προειδοποίηση. Δεν είναι ιδεολογική συζήτηση, είναι τεχνική μαθηματικώς ε, μιλώντας δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο και από πλευράς ποσοτικών και ποσοτικοποιημένων μέτρων είναι πολύ πιο δύσκολο και πιο αβέβαιο. Δεν νομίζω ότι είναι σωστός τρόπος να κινηθούμε προς τα εμπρός. Συνήθως όταν οι παρελθούσες επιδόσεις ε, είναι κακές, ε, ε, το προϊόν μπαίνει σε κάποιο ράφι και χάνεται τελικά, βγαίνει από την αγορά, για να μην φανούν οι κακές παρελθούσες του επιδόσεις. Οπότε θα πρέπει να το δείτε αυτό, γιατί δεν αρκεί. Τώρα για το RTS... Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Για τις συζητήσεις και τις προτάσεις, αυτό είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε από τεχνική σκοπιάς. Είμαι υπέρ δηλαδή της διαδικασίας, μια προσωρινή εξαίρεση. Όμως, σαφέστατα οι ΟΣΕΚΑ πρέπει να συμπεριληφθούν. Και αυτός ο τρόπος ενημέρωσης και πληροφόρησης θα πρέπει να είναι και ο καθημερινότητα, ο κλασικός τρόπος δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τους κανονισμούς και τελικά να καταλήξουμε με ένα μοντέλο που να μην λειτουργεί και να μην είναι έγκυρο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε τη ΣΕΡΠΑ. Επόμενο συνάδελφο από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, δεν βλέπω κάποιον εδώ. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, πάμε στου φιλελεύθερου. Η κυρία Βέρνικε που μόλις έφτασε, που συγκεντρώνεται και ετοιμάζεται για να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Είστε έτοιμοι? Ναι, είμαι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σε ποιο βαθμό η συμπερίληψη των δεδομένων που αποκαλύπτονται συνεπία του, ΠΡΙΠΣ του θα συμβάλλει και θα έχει αντίκτυπο στη ε, θετικό ή αρνητικό στις μελλοντικέ αξιολογήσεις αυτών των προϊόντων και θα επηρεάσει ε, τις εκθέσεις ε, για το κόστος και τις επιδόσεις όλων αυτών των πρίψ. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλεί κανείς από αυτή την επανεξέταση ε, της κατάστασης που επικρατεί σε σχέση με τα πρίψ. Ευχαριστώ. Πράγματι, πολύ συγκεκριμένο το ερώτημά σας. Ευχαριστώ. Έρχομαι στους πράσινους, Βεν Κίγκολτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ με πολλά από όσα ήδη υπόθηκαν εδώ και κυρίως με αυτά που είπε η Σέρπα για το θέμα των παρελθουσών επιδόσεων. Αν ρωτήσουμε τα εμπλεκόμενα μέρη και τους μετόχους που τελικά έχουν συμφέρον να μπουν αυτά τα δεδομένα στο πρίψο, στο πλαίσιο διαβούλευσης, δεν με εκπλήσει που αυτή είναι η απάντηση που παίρνετε και αυτό είναι το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγεται. Εάν οι επαγγελματίες επενδυτές ε, έχουν λόγο, βεβαίω ενδιαφέρονται να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Αλλά εμείς εδώ βάζουμε κανόνες και έχουμε τους επενδυτές λιανικής. Αυτοί πρέπει να μας απασχολούν και να είναι η κύρια μέρημνά μας και το κύριο μέλημά μας. Ακόμα και αν μπει προειδοποίηση ότι οι παρελθούσες επιδόσεις δεν μπορούν να σχετίζονται με τις ε, μελλοντικές. Η συμπεριφορική πλευρά της οικονομικής επιστήμης των οικονομικών μας εξηγεί τι θα κάνει ένας ε, ε, ε, καθημερινός άνθρωπος, ότι δηλαδή θα δει τις παρελθούσες καλές επιδόσεις και θα ελπίσει ότι θα ξανασυμβούν. Τα προϊόντα με κακές επιδόσεις απλά δεν θα του προσφερθούν, ε, ενώ αυτά που έχουν καλές επιδόσεις θα συνεχίσουν να μαρκετάρονται, να μπαίνουν στην αγορά. Και αυτό είναι το κλασικό παραδοσιακό υλικό μάρκετινγκ και... Ε, όμως αυτό δεν είναι μόνο αυτό, είναι δημόσια πληροφορία. Δηλαδή, εμεί πρέπει να περάσουμε το εξής μήνυμα. Εάν επενδύσετε σε προϊόντα, των οποίων η αξία είναι άγνωστη, μη δίνετε πληροφορίες που συντείνουν προς μια αρχή βεβαιότητα. Υπάρχει καλό και κακό σενάριο και υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των πληροφοριών γιατί δείχνουν ότι το μέλλον είναι αβέβαιο. Επομένως, Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, ε, από κοινού Επιτροπή ε, και την Κοινοβουλευτική να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους το γεγονός ότι οι θεσμικοί επενδυτές μπορεί να θέλουν να έχουν πρόσβαση στις παρελθούσες επιδόσεις και καλώς να την έχουν την πρόσβαση αυτή σε, αυτά τα στοιχεία που να βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων, αλλά δεν θα πρέπει οι επιδόσεις αυτές οι παρελθούσες να είναι στο πληροφορικό υλικό, γιατί φαίνεται σαν να είναι δημόσια εγγύηση αυτό, ενώ δεν είναι. Πρέπει δηλαδή ένας θεσμικός επενδυτής να έχει πρόσβαση στο ιστορικό και στις παρελθούσες επιδόσεις του οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικού προϊόντος, αλλά δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται αυτό με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνει εσφαλμένα ή με μη στατιστικός αποδεκτό τρόπο τους ιδιώτες επενδυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Σφέν. Η Γκουέ δεν βλέπω. Η ευθυντή Θα πάρει κάποιος το λόγο. Άλλοι συνάδελφοι. Άλλες παρατηρήσεις, ερωτήσεις παρακαλώ από άλλους ευρωβουλευτές της ΕΚΟΝ. Όχι. Τότε. Να ζητήσω και από τον Καμπριέλ και από τον Σβέ να απαντήσουν παρακαλώ. Αλλά και εγώ έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, είπε η υπερβάωση κάτι πολύ σημαντικό. Εάν η Ένωση Κεφαλαιογορών μπορεί να σημαίνει κάτι για τους επενδυτές, κυρίως για τους ιδιώτες επενδυτές, πρέπει να φτιάξουμε μια πραγματική κεφαλαϊκή ένωση. Ο τρόπος που διαδίδεται η ενημέρωση φυσικά είναι ζωτική σημασία. Δεύτερον, μια κοινή προσέγγιση έτσι ώστε διασυνοριακά η αγορά να λειτουργεί καλά, χρειάζεται μια κοινή θέση. Και αυτό είναι καλό και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση διασυνοριακά για τις εταιρείε. Άρα χρειάζεται μια κατάλληλη και καταναλογία απάντηση στα ζητήματα και η πληροφορία να είναι στοχευμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσει για το προσπέκτους, για τα δείγματα, ο τρόπος με τον οποίο καλύπτονται οι ιδιώτες επενδυτές, το χρονοδιάγραμμα, πώς θα λυθεί αυτό. Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που ακούστηκαν έτσι, πώς θα γίνεται διαβούλευση με τους χρήστες και το ETS. Οπότε παρακαλώ πρώτο κύριος Μπερναντίνο και μετά η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που κάνατε. Θα τα λάβουμε υπόψη μας. Αλλά θα ήθελα τώρα επιτρέψτε μου να καλύψω κάποια σημεία. Πρώτον, για το θέμα της ε, καλύτερης επίδοσης που είναι πολύ σημαντικό. Εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος γι' αυτό. Στη διαβούλευση που κάναμε μια στιγμή διακόπτει ο Πρόεδρος, μια στιγμή. Σας παρακαλώ συνάδελφοι που μπαίνετε στην αίθουσα, το λόγο έχει ο κύριο Μπερναντίνο, οπότε σας παρακαλώ ησυχία. Αν θέλετε να τα λέτε μεταξύ σα, εκτός αιθούση. Κύριε Μπερναντίνο, σας ακούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τις βέλτιστες ε, επιδόσεις. Η θέση μας είναι σαφής. Και Σβέν, για αυτό που είπε και εσύ, δεν είναι μόνο οι ενδιαφερόμενοι φυσικά και ξέρουμε τι θα πει ο κλάδος, εννοείται να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα. και καταλαβαίνω πολλά από αυτά που είπε και εσύ για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Όμως ήταν σαφές από τι απαντήσει που πήραμε από οργανώσεις καταναλωτών, από τους ιδιώτε επενδυτέ, ότι την καλύτερη επίδοση τη βλέπουν σαν τον μοναδικό στόχο. Οπότε θα το κοιτάξουμε. Εγώ προσωπικά Πιστεύω ότι η ενημέρωση για την βέλτιστη επίδοση, αν είναι τυποποιημένη, αν είναι αντικειμενική και με συνοχή, νομίζω ότι είναι μια καλή πληροφορία. Και πρέπει να τη δίνουμε φυσικά με τις ε, ανάλογες ε, ρήτρε επιφύλαξης, έτσι. Ξέρω ότι δεν συμφωνείτε, αλλά γι' αυτό είναι καλή η συζήτηση. Δεν υπάρχει μεθοδολογία για τις μελλοντικέ προπτικές επιδόσεων. Δεν υπάρχει μεθοδολογία που μπορεί να κάνει τέλειες προβλέψεις για το μέλλον. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε και σήμερα με τις ε, δημοσιοποίησεις που κάνουμε. Κάτι μπορούμε να κάνουμε ουσιώδες για τους καταναλωτές να κάνουμε δοκιμές και να δούμε ο κόσμος τελικά τι χρησιμοποιεί από αυτές τις πληροφορίες. Και κάτι άλλο για τη χρήση της εξαίρεσης. Συμφωνώ με το περισσότερα από αυτά που λέει η και άλλοι. Φυσικά τα κενά αυτά πρέπει να καλυφθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί δεν είναι μόνο για του καταναλωτέ, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να καταλάβουν αν υπάρχουν διαφορετικά έγγραφα, αλλά πρόκειται και για την ισοτιμία μεταξύ των χρηστών. Τα PIPs θέλουν να προωθήσουν εξίσου όλα τα προϊόντα και το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα έχουμε τα περί ασφάλειας που συμμετέχουν ενώ τα αμοιβαία δεν συμμετέχουν οι αμοιβές ασφαλίσεις. Κάτι άλλο τώρα για το επίπεδο 2. Η μείωση στην απόδοση. Εμείς καταλαβαίνουμε από τους καταναλωτές ότι δύσκολα μπορούν να το καταλάβουν, οπότε θα δουλέψουμε παραπάνω πάνω σε αυτό το στοιχείο. Και για τα κόστη, το κόστος συναλλαγών, η μεθοδολογία φαίνεται να δίνει κάποιες αρνητικές τιμές. Δεν είμαστε ακόμα πεπισμένοι ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας καλής εφαρμογής της μεθοδολογίας, αλλά ίσως μπορεί και εκεί να υπάρξει κάποια μικρή βελτίωση για περιουσιακά στοιχεία τα οποία να μην έχουν τέτοια ρευστότητα στην αγορά και να μπορεί να γίνει κάποια διόρθωση. Για το SG ε, Pervance, για αυτά που είπες, γι' αυτό φυσικά είναι κάτι σημαντικό εδώ. Τώρα, αν ένας προμηθευτής δίνει ένα στόχο τύπου ESG, αυτό πρέπει να αναφέρεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών, στο KID. Γι' αυτό και εμείς λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιείτε. Ξέρω ότι θέλει πιο συνολικά να το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δικιά μου θέση είναι ότι η δουλειά που γίνεται σήμερα για την ταξινόμηση, η δουλειά που γίνεται επίσης για την επισήμανση στη, στον τίτλο, στις ετικέτες των ε, προϊόντων, πρέπει να κάνουμε κάτι απλό, με χρώματα, με γράμματα, δεν ξέρω, κάτι που να καταλαβαίνει εύκολα ο καταναλωτής. Τέλος, για το θέμα του CMU και τους ιδιώτες επενδυτές. Συμφωνώ, Μπράιν, απόλυτα μαζί Σα, ναι. Αν θέλουμε να έχουμε μια κεφαλαϊκή ένωση στην Ευρώπη σε βάθο, αυτό θα γίνει με του καταναλωτέ. και όχι μόνο με τους επενδυτέ. και γι' αυτό και πιέζουμε για το ΠΕΠ και χαίρομαι που υπάρχει. Και εμεί σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ένα kit και για το ΠΕΠ που είναι διαμορφωμένο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο προϊόν αυτό. Γιατί η δυσκολία που έχουμε είναι ότι έχουμε πολλά διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα, βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και γι' αυτό χρειάζονται διαφορετικές πληροφορίες στους καταναλωτές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις για να είναι πιο εύκολη η συγκρισιμότητα. Ευχαριστώ. Γκαμπριέλ. για να απαντήσει επίσης. Ναι, ευχαριστώ και πολύ σύντομα γιατί δεν νομίζω ότι έχω πολλά να προσθέσω. Το ίσιο, όπως εξηγήσαμε, πρέπει πιστεύουμε να προχωρήσουμε βήμα το βήμα. Έχουμε κάνει προτάσεις για τις πληροφορίες προς κοινοποίηση. Κάνουμε τη δουλειά που χρειάζεται. Ήδη θεωρούμε ότι είναι αρκετές οι πληροφορίες ε, μέσα στο kit. Και δεν χρειάζεται επικάλυψη που άλλωστε δεν θα ήταν και χρήσιμη. Μια συνολική επισκόπηση της νομοθεσίας. Βεβαίως, αυτό θέλουμε να το κάνουμε. Πρέπει να δούμε τι είδους πληροφορίες θα διατίθενται. Με τα προσπέκτους, με το kit, με όλα αυτά. Αρκεί το σύστημα να είναι αποτελεσματικό. Κανένα από τα στοιχεία δεν πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένο. Αυτό επιδιώκουμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Αλλά βέβαια δυστυχώ όπως πάντα, χρειάζεται και το χρόνο του. Κοινοποίηση για κόστο και επιδόσεις. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει. Το είδαμε ιδιαίτερα στο χώρο των ε, ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων υπάρχουν προβλήματα ενημέρωσης, υπάρχει ενημέρωση. άρα πρέπει να κάνουμε κάτι, αλλά με κάποιο τρόπο και να συλλέξουμε την πληροφορία και να την δρομολογήσουμε όπως πρέπει. Πάντως είναι στίγμα του ότι δεν υπάρχουν οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή στα χέρια μας για προηγούμενες επιδόσεις. Πρέπει οι υποπτικέ αρχέ να δουν τι τεχνικέ λύσει μπορούν να δώσουν. Να δώσουν στο επίπεδο 1. Δεν επιτρέπεται να δοθεί πληροφόρηση η οποία θα στηρίζεται μόνο σε προηγούμενε επιδόσει. Μπορεί να υπάρχει ένα μείγμα, μπορεί να υπάρχει διαφορετική λύση. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει σαφή προειδοποίηση. Και εμεί φρονούμε ότι πρέπει να είναι η, ο μορφότυπος ενιαίος για όλους. Για όλα τα προϊόντα, όχι διαφορετικός για κάθε προϊόν, γιατί αυτό θα υπονόμευε τον ίδιο το στόχο που επιδιώκουμε. Άρα δεν πρέπει να γίνει αυτό. Καλώς, ευχαριστώ. Γκάμπριελ, ευχαριστώ Σβέν. Εποπτικές αρχές. και ελπίζω να αποκομίσουμε και τα δάγματα του παρελθόντος. Από τα όσα έχουμε δει και με το kit στο προηγούμενο διάστημα, στα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση σήμερα. Σε ένα λεπτό αγαπητοί συνάδελφοι ξεκινούμε τις ψηφοφορίες. Ας μαζευτούν οι ομάδες, ας οργανωθούν και μόνο για την ΕΚΟΝ, για τις πρώτες ψηφοφορίες είναι μόνο για την ΕΚΟΝ πριν ε, συνεχίσουμε μαζί με τους αδελφούς των προϋπολογισμών. So, let's go to a test. Let's go to a test. Uh, the... Αρχίζουμε δοκιμή. Αρχίζουμε με τη δοκιμή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, παρακαλώ. Μόνο έκον παρακαλώ, όχι μπουτζ. Oh yeah, but I mean, that's always the position. So how are we on numbers? Πώς είμαστε από νούμερα? So we're going to close the vote. Πέρας. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Καλώς. Τέσσερις προφορίες για την ε, οικονομική. Διαδικασίες για μία κέρση αντιρρήσεων. Έμιρ. Παράγραφοι 1 και 2. Παρακαλώ να τις ψηφίσουμε μαζί, αν δεν έχετε αντίρρηση. Παράγραφοι 1 και 2. Ομού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορές 9 7. Ομού. Αν δεν έχετε αντίρρηση. Καλώς. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται αιτιολογικές σκέψεις α και β ομού. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνολικό, συνολική ψηφοφορία για το ψήφισμα. Ονομαστική παρακαλώ. Αρχίζουμε. Πέρασε. Σαράντα υπέρ καμία ψήφο κατά, πέντε απόχέ. Και τώρα έχουμε την έγκαιρη διατύπωση αντιρρήσεων. Πρώτο πρώτος παρακαλώ, υπέρ κατά. Άποχες και εγκρίνονται. Αιτιολογική αναφορά 1 ω 7, εάν δεν έχετε αντίρρηση υπέρ κατά. Όλες μαζί μέχρι το 7 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται αιτιολογικές σκέψεις α και β on block καλό υπέρ και την αιτιολογική σκέψη β, υπέρ κατά υπέρ κατά είναι υπέρ μάλιστα Αποχές και εγκρίνεται και το σύνολο του ψηφίσματος Αρχίζουμε. Να βγει μία ή δύο ψήφοι του ΕΛΚ για τα υπεραριθμούς παρακαλώ. Εντάξει τώρα. Σαράντα υπέρ, καμία ψήφος κατά, έξι εποχές. Τρίτη διαδικασία. Παραγραφή 1 και 2 ομού υπέρ. Όχι, το ΜΑΡ. Η ίδια διαδικασία είναι. Όπως και να έχει. Παράγραφη 1 και 2 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορές 9 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Αιτιολογικές σκέψη α και β ομπλοκ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται και τελική ψηφοφορία ονομαστικά. Αρχίζουμε. Ένας από το L, δύο από το L υπεράριθμοι. Πολύ ωραία. Πέρας. 45 υπέρ. Καμία ψήφος κατά. 7 αποχές. Τελική. Μύφυρ. Παράγραφη 1 και 2 μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές και εγκρίνονται. Τελογικές αναφορές 1 ως 7. Ομπλοκ υπέρ. Κατά. Αποχές και εγκρίνονται αιτιολογικές σκέψεις α και β μαζί, υπέρ, κατά αποχές και εγκρίνονται. Ονομαστικά η τελική ψηφοφορία. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Τι ώρα πράγμα αυτή η συμμετοχή. Πέρας. 45 υπέρ καμία ψήφο κατά, έξι εποχέ και ευχαριστώ του συναδέλφου τη Οικονομικής Επιτροπή για τη συνεργασία. Ένα λεπτό διακοπή για να μπουν και οι λοιποί συνάδελφοι από την Επιτροπή των Αναφυτών Προϋπολογισμών και να συνεχίσουμε με την επόμενη ψηφοφορία.